Θα ήθελα να κάνω μια δήλωση για τα θύματα της τρομοκρατίας στη Βόρεια Ιρλανδία. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η πέμπτη φορά που εορτάζουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα των θυμάτων της τρομοκρατίας. Είναι μια στιγμή μνήμης για τα άτομα τα οποία υπήρξαν αθώα θύματα της τρομοκρατίας. Ήδη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν δύο στρατιώτες στη Βόρεια Ιρλανδία που έπεσαν θύματα του πραγματικού Ήρα, όπως αναφέρεται, και δολοφονήθηκαν. Ο αστυνομικό, επίση, ο οποίο δολοφονήθηκε προχθέ, ήταν παντρεμένο με παιδιά. Η πράξη αυτή της τρομοκρατία έχει και πάλι καταστρέψει μια οικογένεια και έχει φέρει οδύνη σε όλους τους οικείους του φωνευθέντος. Επίσης, υπήρξαν πάνω από 20 άτομα τα οποία σκοτώθηκαν στην Σρι Λάνκα και άλλα τόσα άτομα βρισκόνται μεταξύ ζωής και θανάτου. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να εκφράσω την αγανάκτησή μου για αυτή την αποτρόπη, αυτές τις αποτρόπιες ενέργειες εναντίον αθώων ανθρώπων και να εκφράσω τη συμπαράσταση στις οικογένειες των φωνευθέντων. Θα πρέπει να παραμείνουν όλοι αυτοί στη μνήμη μας. Σήμερα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει στεναρά να εκφραστούμε ενάντια στην τυφλή βία της τρομοκρατίας και καταδικάζουμε απερίφραστα την χωρίς νόημα φώνευση ανθρώπων που είναι αθώοι και που οδηγεί τις οικογένειές τους στην Οδύνη. Μέσα από μία τυφλή αντιμετώπιση η οποία παραβιάζει και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις αρχές της ελευθερίας. Είναι μια παραβίαση της δημοκρατίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας η τρομοκρατία. Είναι η προσπάθεια με την τυφλή βία να καταστραφούν οι αρχές επί των οποίων εδράζεται η, η κοινωνία μας. Πρέπει λοιπόν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη μας να αναχαιτήσουμε τον, την τρομοκρατία. Μόνο με τη στεναρή μας δράση μπορούμε να εμποδίσουμε την τρομοκρατία να υποσκάψει τα θεμέλια των δημοκρατικών κοινωνιών μα. Είναι ένα έγκλημα η τρομοκρατία, κυρίε και κύριοι. Δεν μπορεί να υπάρχει κανένα ελαφρυντικό για την τρομοκρατία. Η τρομοκρατία είναι ένα από τι μεγαλύτερε απειλέ για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τι δημοκρατικέ αξίε τη διεθνού κοινότητα. Είναι μια άμεση επίθεση εναντίον των πολιτών μα και εναντίον όλων μα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και υποστηρίζει τα θύματα της τρομοκρατίας. Δεν μπορούμε να τονίσουμε αρκετά ότι δεν υπάρχει καμία δυνατή αιτιολόγηση και δικαιολογία για τις τρομοκρατικές ενέργειες. Πρέπει οποιοδήποτε αγώνας κατά της τρομοκρατίας όμως να γίνει μέσα στα πλαίσια του κράτους δικαίου και όπως προβλέπει ο νόμος στις χώρες μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει και πάλι την ενθύμησή του και την συμπαράστασή του με όλα τα θύματα της τρομοκρατίας όπου να ζουν όπου να ζούσαν στον κόσμο μας. Για να σε, σε ένδειξη τιμής προς τα θύματα του Ήρα και στο, στα θύματα του Σιλάνκα σας ζητώ να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από 30 χρόνια, στις 16 Μαΐου του 1979, ο Ζαν Μονέ, ένας από τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πνευματικός πατέρας της, απέθανε. Με την ευκαιρία αυτής της επαιτίου θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή την ε, συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέροντας το έργο του Ζαν Μονέ για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα ενθυμούμαστε την εξαιρετική συμβολή ενός ανθρώπου ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει την συμφιλίωση μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας που ήταν το πρώτο βήμα για μια ειρηνική συνεργασία σε ένα κοινό ευρωπαϊκό χώρο που επεκτάθηκε στη συνέχεια σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα, μέσα στον 21ο αιώνα, είναι πολύ σημαντική η συμβολή του Ζαν Μονέ και η μέθοδος την οποία ακολούθησε τότε πριν από 50 χρόνια δεν έχει χάσει καθόλου την επικαιρότητά της. Μπροστά στις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική κρίση, με την αλλαγή του κλίματος, θα πρέπει η Ευρώπη όλο και περισσότερο να συνεργάζεται να συνεργάζονται τα κράτη της Ευρώπης πιο στενά και να μπορέσουν να τηρήσουν και να διατηρήσουν τις αξίες τους στο διεθνές στίβο. Ο Ζαν Μονέ έχει βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας και της πολιτικής ένωσης. Και αυτά θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να κάνουμε και εμείς τις προσπάθειες να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στον 20ο αιώνα που να είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Και αυτό μας ενθυμίζει ότι ο Ζαν Μονέ είχε ονειρευτεί και τις άμεσες εκλογές της ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό έγινε πραγματικά πραγματικότητα μετά το θάνατο του Ζαν Μονέ με την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε όλοι κληρονόμοι αυτού του μεγάλου Ευρωπαίου του Ζαν Μονέ. Το έργο του είναι διαρκές και αέναο και η επιρροή του εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και σήμερα για όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ευκαιρία λοιπόν των 30 ετών από το θάνατο του Ζαν Μονέ, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα καθήκοντα που έχουμε προς το μέλλον να συνεχίσουμε το έργο του Ζαν Μονέ το οποίο θα οδηγήσει στην πραγματική ένωση της Υπήρου μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Κομισιόν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Θεωρούμε ότι το σύνολο της